που συμπεριλαμβάνεται. Όλη η βοήθεια του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ κυρία Ρέντινγκ. Τελειώσαμε με το θέμα αυτό και η ψηφοφορία θα γίνει πραγματικά αύριο αυτή τη φορά.